Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Μαρτελή, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ΑΕΤ, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικές. Ο σοβαρός σεισμός της 12 η Ιανουαρίου 2010 ο οποίος συγκλώνησε την ΑΕΤ και ε, οδήγησε θάνατο πάνω από 220.000 ανθρώπους και έκανε αστέγους 1,7 εκατομμύριο άλλους επέφερε μια διεθνή αλληλεγγύη και πρωτοφανή κινητοποίηση κυρίως των Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανθρωπιστική βοήθεια ευρεία κλίμακα και ε, αναπτυξιακή βοήθεια για την ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση τη χώρα σα. Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερο δωρητή στην παροχή βοήθεια για την ΑΕΤ. Ενώ η χώρα σας αγωνίζεται ακόμα να ξεπεράσει ε, τις ολέθριες συνέπειες του σεισμού, ε, φέτος επλήγει για δεύτερη φορά από μια θεομηνία θεομηνίες ε, οι κυκλώνες Ισακ και Σάντι και πάλι έφεραν τον όλεθρο και την οδύνη στη χώρα με καταστροφικές συνέπειες ε, στην παροχή βοήθεια στον πληθυσμό. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, αγαπητέ κύριε Μαρτέλη, το κοινοβούλιο μας ανέκαθεν αγωνίζονταν για ε, ισχυρή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΑΕΤ και στενή συνεργασία με τις αρχές της χώρας. Θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα σας. Επιθυμούμε να βοηθήσουμε για μια IT ε, ε, ε, που να είναι οικονομικά και πολιτικά σταθερή και θα μπορεί να αναλάβει τις τύχες της και να μπορεί να συνεισφέρει και ίδια στην προσπάθεια της βιώσιμης μείωσης της ένδυας. Στο πρόσωπό σας ε, βλέπουμε ε, την ελπίδα για εγκαθίδρυση σταθερής δημοκρατίας και βιώσιμης στην ΑΕΤ. Οι προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαρτέλη είναι τεράστιες και πιστέψτε μας γνωρίζουμε, αυτό άλλωστε το έδειξε και η χθεσινή συζήτηση στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές Γνωρίζουμε πόσο δραματικές είναι αυτές οι προκλήσεις. Τρία έτη μετά την καταστροφή περιμένουν ακόμα 370.000 πολίτες ε, να στεγαστούν με τρόπο αξιοπρεπή γιατί σήμερα ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες και είναι πάρα πολύ σημαντική ε, η βοήθεια που χρειάζεται η διαδικασία ανοικοδόμησης. θα πρέπει λογικά να ε, διαμορφωθεί όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά η ένδυα στη χώρα να καταπολεμηθεί με κάθε μέσο και η ενίσχυση της δημοκρατίας που είναι τόσο απαραίτητη και του κράτους δικαίου χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Ειδικά η δικαιοσύνη είναι ένα θέμα που πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί. Και θα ήθελα να προσθέσω εν ώψη της συζήτησης για τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και στο μέλλον στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Ακριβώς απέναντι στη δική σας χώρα. Θα πρέπει εμείς να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και να δείξουμε στους πολίτες της ΑΕΤ, άνδρες και γυναίκες, ότι είμαστε συμπαραστάτες στο πλευρό τους με αλληλεγγύη. Για να μπορέσετε εσείς να εφαρμόσετε το δικό σας φιλόδοξο ε, πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο είναι στο πλευρό σας και θα αγωνιστεί ε, για να ε, εξασφαλίσει τα κονδύλια που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τηρήσει τις υποχρεώσεις και απέναντι στην ΑΕΤ. Εξού και ο αγώνας μας για ένα φιλόδοξο κοινοτικό προπολογισμό είναι και ένας αγώνας για την εγγύηση ότι τηρούμε τις υποσχέσεις μας για τη διεθνή ελληνική. Έχω τώρα τη ε, χαρά, κύριε Πρόεδρε τη Δημοκρατία, να σας δώσω το λόγο και σας καλωσορίζω και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, είναι ιδιαίτερη η τιμή που κάνετε στη χώρα μου με την υποδοχή μου εδώ στο περίβλεπτο Κοινοβούλιο του Στρασβούργου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, έρχομαι εδώ κομίζοντας ένα άλλο πιστεύω. Το ίδιο πιστεύω που σας ενέπνευσε στους χαλεπούς καιρούς. Το ίδιο πιστεύω που σας επέτρεψε να ζήσετε τα 30 χρόνια της Μεγάλης Ευμάριας. Το ίδιο που σας επέτρεψε να ορθοποδήσετε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ίδιο πιστεύω που έριξε το τείχος του Βερολίνου. Το ίδιο που εμψύχωσε τον αξιοσέβαστο Πόλαν Ρισπακ. Έρχομαι εδώ για να σας διαμηνήσω ότι παρά τις αντικσοότητες, παρά τις ταλαιπωρίες και τα βάσανα, η ΑΕΤ δεν υπέκυψε. Αργά, αλλά σταθερά, η ΑΕΤ συνέρχεται. Και αυτή τη χαρμόσυνη είδηση ήθελα να σας μεταφέρω εδώ. Αυτή η αλλαγή πορείας που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο θάρρος του λαού μας, στην αποφασιστικότητα της διοίκησής μας, ταυτόχρονα οφείλεται και στην δυναμική συνεργασία της Ευρώπης, που είναι η πιο σημαντική από όλες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Βλέπω στη συνεργασία αυτή τα σημάδια μιας φιλίας που σφυριλάτησε η ιστορία Μία φιλία που δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους απέναντι στη χρηματοπιστωτική κρίση που απειλώντας εσάς αγγίζει και εμάς. Είμαι πεπισμένος ότι η Ενωμένη Ευρώπη και άρα πιο ισχυρή Ευρώπη θα καταφέρει να βρει τις κατάλληλες λύσεις για να ανακάμψει και πάλι οικονομικά. Πιστεύω ακράδαντα ότι καμία ύφεση δεν είναι μόνιμη. Η διάρκεια μιας κρίσης εξαρτάται από την ταχύτητα και την ευστοχία των μέτρων ανάκαμψης. Από το Μάριο Ντράγκη μέχρι την Κριστίν Λαγκάρτ, για να αναφέρω μόνο δύο, έχετε μερικά από τα καλύτερα μυαλά του πλανήτη που θα σας επιτρέψουν να τη θασεύσετε την κρίση και να τη διορθώσετε. Αλλά με την παρουσία μου εδώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη γενεοδορία σας και για την αλληλεγγύη σας και να υπενθυμίσω ότι καμία χώρα δεν θα καταφέρει να εξέλθει από τη φτώχεια ζώντας από φιλανθρωπίες. Σίγουρα η ΑΕΤ χρήζει ακόμη αρρωγής, αλλά οι κάτοικοί της Χρειάζονται περισσότερο παραγωγική εργασία. Χρειάζονται εμπορικές συναλλαγές και άμεσες επενδύσεις. Η ΑΕΤ βρίσκεται στις πύλες της Αμερικής. Της Αμερικής του Βορρά που ξαναρχίζει να αναπτύσσεται και της Νότιας Αμερικής που αυτή τη φορά δεν έπεσε σε κρίση και δεν σταμάτησε ποτέ την ανάπτυξή της. Η ΑΕΤ είναι μια πλατφόρμα στρατηγικής σημασίας. Ένα πρόσφορο επενδυτικό κλίμα. Ένα εφαλτήριο που μπορεί να επιτρέψει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην ανοικοδόμησή της και ταυτόχρονα να έχουν ένα σημαντικό προπύργιο για την περιοχή. Η ΑΕΤ χρειάζεται λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμους, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρειάζεται ξενοδοχεία. Η Αιτή έχει ένα γόνιμο έδαφο και μπορεί εύκολα να ξαναρχίσει να θρέφει τον πληθυσμό τη και να εξαγάγει τα πλεονάσματά τη. Η Αιτή έχει ένα παρά, απαράμιλο κλίμα και γεωγραφία. Χιλιάδες χιλιόμετρα παραλίες με λευκή άμμο και μια φύση που σε μεγάλο βαθμό έχει μείνει παρθένα και ανεξερεύνητη. Από το Φόρτ Λιμπερτέ μέχρι τη Σκάγια, από την Κοναΐβ μέχρι τη Μυραγκουάν, η χώρα μας βρήθη φυσικών λιμανιών με βαθιά νερά. Ο πληθυσμός μας είναι νέος, γενναίος, προσινής, εργατικός. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω, να σας προσκαλέσω και να σας παρενέσω να αξιοποιήσετε στο έπακρο το δυναμικό της χώρας μου και τις καταπληκτικές επενδυτικές της ευκαιρίες. Σας προσκαλώ να συνεργαστείτε μαζί μας για να μας βοηθήσετε να ξανακατακτήσουμε τη χρηματοπιστωτική μας κυριαρχία για να μπορέσουμε να, να επιστρέψουμε στις διεθνείς χρηματαγορές. Βρίσκομαι εδώ ώστε από κοινού να εξετάσουμε νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Σας παροτρύνω να συνεργαστούμε για να σχεδιαστούμε και να δρομολογήσουμε έξυπνα και αποδοτικά προγράμματα. Σας ζητώ τη συνεργασία σας για να μπορέσουμε να βρούμε από κοινού τα καλύτερα προγράμματα για τη χρηματοδότησή τους. Πολλοί από τους συνταξιούχους καθηγητές σας ονειρεύονται να συμβάλλουν ώστε να γίνει ο κόσμος μας πιο δίκαιος. Στείλτε τους εμάς για να συμμετέχουν στην επιμόρφωση των νέων μας και των δικών τους δασκάλων. Μπορείτε έτσι να συμβάλλετε ώστε να αλλάξουμε μαζί την ιστορία. Η ιστορία που μας υπενθυμίσει τους δεσμούς μας με την Ισπανία, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία. Η πιο πρόσφατη ιστορία που μας παραπέμπει στις εμπορικές μας σχέσεις με τη Γερμανία πριν το 1940. Η ιστορία που επίσης θα συγκρατήσει αυτό που κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τις προσπάθειές της για αναπτυξιακή συνεργασία. Η Ευρώπη μπορεί να είναι υπερήφανη για τη θέση που έχει στον κόσμο, για το χάρισμά της, τις πεπιθήσεις της, τις ιδέες της, τις λύσεις που δίνει στα προβλήματα του πλανήτη, τις πρωτοβουλίες της, και το ρόλο της στις αναδυόμενες χώρες. Η ευρωπαϊκή νεολαία πρέπει να γνωρίζει ότι οι χώρες του Νότου περιμένουν πολλά από αυτήν. Δεν μπορεί να παραμείνει εσωστρεφής. Από τη γενναιοδορία και τις έξυπνες επιλογές της ε, θα προκύψει ένας κόσμος με μεγαλύτερη αδελφικότητα, πιο ηθικός οικονομικά, πιο ασφαλής οικολογικά σίγουρα πιο δυναμικός, πιο δημοκρατικός και πιο ανεκτικός. Η ΑΕΤ σήμερα, ισχυρή με την φιλή αυτή, αρχίζει και συνέρχεται, διαγράφει τα παλιά στερεότυπα, διαρριγνύει τις, αλη... τις αλυσίδες της ενδημικής υποανάπτυξης, εξορκίζει τους παλιούς τις δαίμονες, δίνει μάχη κατά της απερίμωσης που την απειλεί και θέλει να ανοίξει προς τον κόσμο. Εδώ και ένα μισή χρόνο με αυτό ασχολείται η, η δημόσια διοίκησή μας. Με αδεξιότητες μερικές φορές, αλλά κανένας δεν μπορεί να αφιβάλλει για το ότι είμαστε καλοπροαίρετοι. Φέτος ακόμη, η IT επλήγει με διαφορετική ένταση από τις τροπικές καταιγίδες Ισάκ και Σάντι. Μία ακόμη φορά είχαμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, σε σοδιές, σε κατοικίες, σε ζώα. Μία ακόμη φορά η διεθνής κοινότητα έσπεψε να μας συνδράμει, να διασώσει, να ανοικοδομήσει. Κάποια μέρα θα πρέπει να διαρρήξουμε αυτό το φαύλο κύκλο και να φτιάξουμε έναν ενάρετο κύκλο αυτό επιδιώκουμε. Και χάρη σε αυτές τις προσπάθειες θα ορθοποδήσει και πάλι η ΑΕΤ. Η ΑΕΤ θα ανασυγκροτηθεί γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο ευάλωτο είναι το έδαφος μας. Και μάλιστα η κατάσταση αυτή θα, επιδεινωθεί στο μέλλον, στο μέτρο που εντείνονται οι κλιματικές αλλαγές που έχουν αναγγελθεί για τις αντίλες. Η ΑΕΤ όμως θα ορθοποδήσει γιατί πεισματικά ασχολούμαστε και με ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό στον χρόνο, το θέμα της πρόληψης. Και η πρόληψη στον τομέα αυτό έχει το όνομα της χωροταξίας. Με τη χωροταξία θα καταστήσουμε τη χώρα μας λιγότερο ευάλωτη. Θα προστατεύσουμε τις λεκάνες απορροής ώστε να σταματήσουν εξαιτία τη αποψήλωσης, της διάβρωσης και της άναρχης δόμησης να γίνονται αιτίες καταστροφής. Χωροταξία σημαίνει να μην χάνουμε σε κάθε θεομηνία χιλιά, εκατομμύρια δολάρια. Χωροταξία σημαίνει να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο αποδεκτό για τον πληθυσμό της αιτής. Η κυβέρνησή μου έχει εργαλεία ώστε να κάνει πραγματικότητα τη χωροταξία. Τα εργαλεία αυτά είναι το Εθνικό Κέντρο της Γεωχωρικής Πληροφόρησης που στηρίζεται από εσά, την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΣΙΑΤ, την Διυπουργική Επιτροπή Χωροταξίας, στην οποία και εσείς συμβάλλετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η διοίκησή μου θα χρησιμοποιήσει στο έπακρο τα εργαλεία αυτά και σε βάθος χρόνου, ώστε να αφήσει το στίγμα της στην επικράτεια της ΑΕΤ και στο έδαφος της. Βλέπετε ότι στον τομέα αυτό η η Ήπειρό σα προηγείται πολλών εταίρων. Όπως λέμε εμεί ε, η Ευρώπη πάει μπροστά. Η γυρά ήπειρο συνεχίζει να είναι πηγή έμπνευση σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου όλο και περισσότερο τα κράτη που ήταν μοναχικοί καβαλάριδες θα πρέπει να δώσουν σε μεγαλύτερη περιφερειοποίηση, να δημιουργήσουν ελεύθερε ζώνε κυκλοφορία αγαθών και προϊόντων, να μιλούν με μια ενιαία φωνή, ε, να αλληλοβοηθούνται, διατηρώντας όμως την ταυτότητά τους. Η περιοχή της Καραϊβικής μαζί με τις μικρές και τις μεγάλες αντίλες μπορεί κάποια μέρα να αναδειχθεί ως πραγματική ένωση ανεξάρτητων κρατών και να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό της καταπληκτικής γεωστρατηγικής της θέσης. Αυτό δεν είναι μόνο το τίμημα της σταθερότητας, θα έλεγα και της ειρήνης στον κόσμο αλλά είναι και κάτι παραπάνω. Είναι τα νέα κίνητρα για την ανάπτυξη σε ένα πλαίσιο όπου όλοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόσουν την ειρήνη και να δεσμευτούν υπέρ της νομοτυπίας και της δικαιοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της συνδρομής της προς τις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού συμβάλλει και μάλιστα τα κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στο κεφάλαιο της περιφερειακής ολοκλήρωσης, τα κονδύλια αυτά αυξάνονται και συμβάλλουν στην πρωτοβουλία που σας περιέγραψα. Η ΑΕΤ σήμερα έχει επίγνωση της θέσης της, του βάρους και του ρόλου της στην περιοχή. Γνωρίζει όμως ταυτόχρονα και τα κενά της. Με διάβγεια αξιολογήσαμε τις καθυστερήσεις μας και χωρίς αυτομαστίγωση προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά και θα τα καλύψουμε. Κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Δεν θα είναι ένας αγώνας ταχύτητες, αλλά ένας αγώνας αντοχής. Και εκεί αντλούμε την έμπνευσή μας από την Ευρώπη. Γιατί αν κάποιες χώρες μέλης της ήταν αθεμαγμένα μόλις πριν από μισό αιώνα, σήμερα και παρά τη χρηματοπιστωτική κρίση στηρίζονται ακόμη σε πολύ γερά θεμέλια που θα τους επιτρέψουν μια μέρα να συνέλθουν και να ορθοποδήσουν. Η ανάκαψη της Ευρώπης εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τη διαφανή διαχείριση των δημοσίων πόρων, από την ορθολογική τους χρήση, από τη σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης, από το μορφωτικό επίπεδο των πληθυσμών από την επιθυμία τους να εργαστούν άοκνα για να ανατάξουν τις οικονομίες τους. Η επιτυχία δεν γνωρίζει σύνορα. Θα αφιερώσω τη θητεία μου μεταξύ άλλων στην παιδεία, στη μόρφωση του πληθυσμού μας, στην πάταξη της διαφθοράς, στην εγκαθίδρυση ενός κράτους δικαίου. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε αποτελέσματα σε αυτή την προσπάθεια. Ήδη πριν από λιγότερο από δύο χρόνια, πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά που μέχρι τότε ήταν εγκαταλελειμμένα, εντάχθηκαν δωρεάν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και μάλιστα αποκλειστικά με δημόσια κονδύλια. Ήδη βλέπουμε την προσπάθεια της ανασυγκρότησης με την παροχή στέγη σε πάνω από ένα εκατομμύριο στέγους, δικαιώνοντας έτσι και τις προσπάθειες που κατέβαλαν και οι δικοί σας φορολογούμενοι. Θα ήθελα να τους εκφράσω την αμέριστη γνωμοσύνη μου και να τους διαβεβαιώσω ότι η αλληλεγγύη τους δεν πήγε χαμένη. Ότι έφτασε στους πιο ευάλωτους Το κράτος δικαίου που επιθυμούμε αρχίζει και παρουσιάζεται με τις εξής μορφές. Με την πλήρωση των θέσεων εργασίας στα θεσμικά μας όργανα. Με την έγκριση της συνταγματικής αναθεώρησης παρά τις αδυναμίες της. Με την αποκατάσταση του δικαστικού σώματος. Με την ορκομοσία του Συνταγματικού Συμβουλίου με τη θέσπιση του μόνιμου εκλογικού συμβουλίου. Με τις επερχόμενες εκλογές που θα ανανεώσουν το 1 τρίτο της γερουσίας μας. Με τις πολιτικές ελευθερίες που ισχύουν. Με την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης και για την αντιπολίτευση. Με την υποχώρηση της διαφθοράς και με τη δίωξη του εγκλήματος που δεν θα βρίσκει πια πουθενά κρυσφύγετο. Αργά αλλά σταθερά η δικαιοσύνη μας γίνεται πιο δίκαιη. Στο κεφάλαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εργάζομαι πυρετοδός προκειμένου να κυρωθούν στη διάρκεια της δικής μου θητείας συμφωνίες και συνθήκες για την ισχύ του απαράγραπτου για ορισμένα εγκλήματα. Στο ίδιο κεφάλαιο, στη διάρκεια της θητείας μου και με τη δική σας συνεργασία, το δικαίωμα στην υγεία, την εργασία, την ισότητα των ευκαιριών, στην ισότητα των δύο φύλων, στην προστασία των ανηλίκων. Όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα. Τα πρώτα σημάδια είναι ήδη αφάνη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, εν αρχή είναι η οικονομική Ευρώπη. Οι ιδρυτές πατέρες της ΕΟΚ το είχαν καταλάβει θα έπρεπε να το καταλάβουν και οι χώρες ΑΚΕ και ιδιαίτερος η ΑΙΤ. Η συνεργασία σας αυτό το σκοπό έχει με την συνδρομή σας σε μείζωνα έργα υποδομής. Η Εθνική Οδός Υπαριθμόδια 2 με τα εγγένεια μεγάλου τμήματός της παρουσία του Επιτρόπου Πίμπαλξ ήταν ένα εύγλωτο σημάδι. Με το δρόμο αυτό, με την οδό αυτό θα ξαναδώσουμε δυναμισμό στις τοπικές οικονομίες και σας είναι ευγνώμονες ε, οι τοπικές οικονομίες γι' αυτό. Τα εργαστήρια μεταποίησης ε, πρώτων υλών στα σύνορα με τους ε, γειτονές μας, τα τελωνία και προσπάθειες απελευθέρωσης των εθνικών αγορών στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και ήδη από την αρχή της θητείας μου τάχθηκα υπέρ όλων αυτών των αρχών και υπέρ πολλών αρχών ακόμη. Των αρχών που πηγάζουν από τη δική σας σοφία, από τα δικά σας ιδανικά και από τον αρχαίγωνο πολιτισμό σας. Τις αρχές που ακτινοβολούν από το Στρασβούργο που συνδέεται πια άρρηκτα με τα δημοκρατικά ιδεώδη του κοινοβουλίου σας. Τις αρχές ε, χάρη στις οποίες μας παραστέκεστε και τις αρχές στο όνομα των οποίων με υποδεχτήκατε σήμερα εδώ με τέτοια συντροφικότητα και οικειότητα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε για τα λόγια σας. Και επίσης, για τις αναφορές σας στους ε, ιδρυτές πατέρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ήταν και για μας η ομιλία σας ενθάρρυνση ε, για να προχωρήσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που είναι σημαντική όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για άλλα μέρη του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ και αγαπητοί συνάδελφοι για την προσοχή σας και σας ευχόμαι καλή επιτυχία για το υπόλοιπο των εργασιών σας. Ευχαριστώ.